Good morning, ladies and gentlemen. We're running slightly late. It's past. Κυρίες και κύριοι, καλό είναι να ξεκινήσουμε. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Είναι 9 και 10. Θέλω να σας καλωσορίσω στην κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ και ΔΕΒΕ για την ανάπτυξη, τη γειτονία και τη διεθνή συνεργασία στο καινούριο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. ότι η ακρόαση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ανάλυσης των προτάσεων της ε, Κομισιόν για, την, για το Μηχανισμό Ανάπτυξης γειτονία και Διεθνούς Συνεργασίας. Σημαντική διαδικασία διότι ε, θα καθορίσει το πώς θα δαπανηθούν τα, τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία προβλέπονται μέχρι το 2027 για βοήθεια σε τρίτες χώρες. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η συνήθις ε, νομοθετική διαδικασία. Αφεντεύε είναι συνυπεύθυνε στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον κανόνα 55. Η πρόταση αυτή είναι λοιπόν σημαντική και γι' αυτό το λόγο έχουν οριστεί τέσσερις συνεισηγητές, δύο και δύο από την κάθε επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται την έκθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Ο στόχος μας σήμερα είναι να αξιολογήσουμε το σε ποιο βαθμό το νέο, ο νέος αυτός μηχανισμός θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι διεθνής παίκτη και να πετύχει τους στόχους της βιώσιμη ε, βιώσιμης ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα έγγραφά σας θα έχετε δει, έχουμε δύο πάνελ. Πρώτον, ανάπτυξη, ε, χρηματοδότηση και ε, συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη μέχρι το 2020 και το δεύτερο πάνελ πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτός ο μηχανισμός θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο αποτελεσματικός παίκτη στη δημόσια σκηνή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρεντς, ο οποίος θα συντονίσει το πρώτο πάνελ, αλλά πριν από αυτό να δώσω το λόγο και στη συμπρόεδρο, την κυρία Μακάβεν. Ε, υπάρχουμε μια ομάδα από την Plan International εδώ. Πού είσαστε? Α, μόλις τώρα μπήκανε. Έχουν έρθει στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή ε, Εβδομάδα Δράση για τις Γυναίκες. Ε, με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας για τις ε, γυναίκες για τα κορίτσια. Μιλάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα χρηματοδοτήσουμε και τέτοιες δράσεις. Ελπίζω θα υπάρχει και μια ισχυρή διάσταση χρηματοδότησης τέτοιων δράσεων για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Oui, merci, monsieur euh, et madame euh, le président. Euh, chers collègues. ξεκινάμε αυτό το πρώτο τμήμα της ε, κρόσης εξετάζοντας την αντισιακή ε, μα πολιτική και τις επιπτώσεις που θα έχει ο καινούριος μηχανισμός επί αυτής. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον μηχανισμό αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Ορισμένα βέβαια θα διευκρινιστούν μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή του κανονισμού. Κάποια άλλα ερωτηματικά μπορούν να διευκρινιστούν ήδη από τώρα και να βελτιώσουμε το κείμενο έτσι ώστε αυτό το, αυτός ο μηχανισμός των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες των τρίτων χωρών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε λοιπόν να δοθούν πολλές διευκρινήσεις σήμερα, ιδιαίτερως να ακούσουμε αυτές και αυτούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του μηχανισμού, δηλαδή τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εξπροσωπούνται σήμερα από την Concord. Η συνοχή των εσωτερικών μας και εξωτερικών μας πολιτικών αφενός και των εξωτερικών μας πολιτικών μεταξύ τους αφετέρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο, ο, ο, ο, ο, θα μας διευκρινίσει το δικό του ρόλο και την άποψή του για αυτό το μηχανισμό και για άλλους υπάρχοντες μηχανισμούς. Καλωσορίζουμε την κυρία Έμπα ε, προϊστάμενη για την ε, συνοχή πολιτικών και για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον ΩΣΑ, καθώς επίσης και την κυρία Άλβα Φιν της οργάνωσης Save the Children, που θα μιλήσει εξ ονόματος της Concord, που είναι η Συνομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ευρώπης για την ακούφιση και την Ανάπτυξη. Δίνω το λόγο σε αυτές τις κυρίες, 7 ε, λεπτά στην καθεμία και ξεκινάμε με την κυρία Έμπα Ντόλμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ομολογήσω ότι όταν με προσεγγίσατε με τον ε, τίτλο της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, ε, σκέφτηκα ότι ο διευθυντής μου θα ήταν ε, πιο κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσει για το θέμα αυτό συζητάμε τις ε, συστάσεις, θα συζητήσουμε μάλλον ε, τις ε, συστάσεις που θα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προκύψουν στις 24 Οκτωβρίου. Ελπίζω να έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι πιο ικανοί συνάδελφοί μου να σας παρουσιάσουν τα θέματα αυτά. Στο μεταξύ όμως χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ να σας μιλήσω για την πολιτική συνοχή και γιατί είναι κατάλληλο εργαλείο για να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, χωρίς να μένει κανένας πίσω. Θα είναι επίσης ε, μια ευκαιρία να τονίσω γιατί είναι τόσο σημαντικό το μέσο γειτονίας ανάπτυξης ε, και διεθνούς συνεργασίας. Όπως πιθανότατα να γνωρίζετε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι αρκετά διαφορετικό πράγμα από τους στόχους της χιλιετίας. Είναι πολύ πιο ευρύ το θεματολόγιο, λαμβάνονται υπόψη η σχέση μεταξύ των διαφόρων στόχων και των διαφόρων διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Διότι για να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση πρέπει να αναγνωριστούν οι διαφορετικές μορφές φτώχειας, για παράδειγμα. Δεύτερον, ε, λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ε, διασυνοριακές επιπτώσεις αλλά και τις διαγενειακές επιπτώσεις και αναγνωρίζεται ότι γίνονται παραχωρήσεις ε, για να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στις, στους τοπικούς στόχους και τους διεθνείς και στους ευραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Υπάρχουν διάφορες ανάγκες που θα πρέπει να ε, καλυφθούν για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το φιλόδοξο θεματολόγιο. Έχουμε λοιπόν έναν ορισμό, διότι νομίζω ότι όλα πρέπει να ξεκινήσουν από ορισμό της προσέγγισης. Λέμε λοιπόν ότι η πολιτική συνοχή για βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση και ένα μέσο πολιτικής ε, που ε, θα βοηθήσει την ε, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα λήψη αποφάσεων και υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Τη βιώσιμη ανάπτυξη Να σας δώσω ε, κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ανταγωνισμό ανάμεσα στους διάφορους στόχους, ο στόχος 7-2 θα μπορούσε ε, να συγκρούεται με τον στόχο 2.1. Ε, μπορεί δηλαδή να έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσα στα βιοκαύσιμα και στα τρόφιμα ή οι ενισχύσεις ε, στα ορυκτά καύσιμα ε, έχουν οικονομικό κόστος, ε, επηρεάζουν τον ανταγωνισμό, επίσης επιφέρουν περιβαλλοντικό κόστος λόγω των εκπομπών και έχουν επίσης και κοινωνικό κόστος, διότι επηρεάζουν την υγεία με την ρήπανση του αέρα, κάτι που μειώνει το προσδόκιμο ζωής. Άλλο παράδειγμα είναι οι χρηματικές ε, ροές, η νομοποίηση παράνομων εσόδων ε, και το υψηλό κόστος συναλλαγών. I think we need to look Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να εξετάσουμε το στοιχείο αυτό των συμβιβασμών που γίνεται ανάμεσα ε, στην ευημερία μας εδώ και τώρα και τις διασυνοριακές επιπτώσεις καθώς και την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων, διότι μπορεί κανεί να επικροτήσει την πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική εμπορίου με στόχο την υποστήριξη φτωχών χωρών ε, με το ε, σύστημα προτιμήσεων και το σύστημα τα πάντα εκτός από όπλα, αλλά ε, βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να εξωτερικεύεται το, οι εκπομπές με τη μετακατάσταση εργοστασίων. Επίσης, ε, οι γεωργικές ενισχύσεις ε, στρεβλώνουν την αγορά. Αναγνωρίζουμε την ε, ανάγκη διασφάλισης της επισητιστικής ασφάλειας. Βλέπουμε όμως και μεγάλη σπατάλη τροφίμων. Και θα πρέπει να το ζυγίσουμε αυτό σε σχέση με Θα πρέπει να ζυγίσουμε την ε, κατανάλωση νερού με την ε, ανάγκη για νερό στην παραγωγή, ε, τη γεωργική παραγωγή. Επίσης, τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα έχει εισαγόμενη σόγια που χρησιμοποιείται και στα τρόφιμα αλλά και ως ζωοτροφή. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να επανέλθω στα μέσα που συζητάμε εδώ πέρα, συγκεκριμένα το NDICA, την πολιτική συνοχή για Το, το μέσο γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Είχε προταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την συνεργασία ε, ευθυγραμμίζοντας ε, τους ε, κανόνες, απλοποιώντας ε, τις γραμμές του υπροπολογισμού και απλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να γίνει η διαδικασία πιο αποτελεσματική και ευέλικτη. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή που εκδόθηκε πρόσφατα επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλους τους τομείς αυτούς. Και το NDICI ε, πράγματι απλοποιεί ε, τη διαδικασία και αυξάνει την ευελιξία. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να διακυβεύσουν τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι η ε, εκρίζωση της φτώχειας. Εξετάζουμε λοιπόν ε, την ε, συνεκτικότητα των πολιτικών σε τέσσερα επίπεδα. Καταρχάς, όσον αφορά τα διάφορα είδη χρηματοδότησης και πιστεύω ότι το μέσο αυτό ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ως προς αυτή την πτυχή, ε, δηλαδή την απλοποίηση των διαδικασιών. Το μέσο αυτό θα είναι πάντα σημαντικό για την εκρίζωση της Φτώχεια ε, και το να υπάρχει συνεκτικότητα ε, θα έχει θετικές επιπτώσεις. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς ε, αν αρκεί και αν λαμβάνει υπόψη και άλλα μέσα για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα κλείσω με ετούτη τη διαφάνεια που ε, δείχνει το πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτικών. Θα κλείσω εδώ και θα ήθελα να ακούσω λεπτομέρειες σχετικά με το μέσο από τους άλλους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame Dolman. J'invite maintenant Madame Alvafine à prendre le relais. Uh, thank you for giving Concord the opportunity to weigh on, in on the Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά μου Αλβίνα και εργάζομαι για την, ε, το Ίδρυμα Save ε, Children και για μια Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδία που αποτελείται από 55 μέλη που εκπροσωπούν πάνω από 2.000 ΜΚΟ. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ένας ξεχωριστός μηχανισμός. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς θα λειτουργήσει νέα αυτή η προσέγγιση, αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τα θετικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Πραγματικά έχουν, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες ε, που προκύπτουν από αυτό το μηχανισμό. Ε, υπάρχει ένα θεματικός πυλώνας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η νέα γεωγραφική προσέγγιση είναι επίσης ευπρόσδεκτη και υπάρχουν ενδείξεις ότι ότι η Ένωση θέλει να αντιμετωπίσει τα ανθρωπιστικά θέματα. Επίσης, ο συνυπολογισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλα αυτά να βρίσκονται στο κέντρο του μηχανισμού. Βεβαίω, υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι το θέμα της ελαστικότητας, τη ευελιξίας έχει κινηθεί, έχει τίνει πολύ προς, προς μία κατεύθυνση. Επίσης έχουμε και άλλους ε, προβληματισμούς. Ελπίζω, αυτό το μηχανισμό συνδυάζει διάφορους τομείς ε, της πολιτικής, αλλά κατά την άποψή μας δεν επιτυχάνει μια ισορροπία μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης, προκειμένου να υπάρχει ένα σωστός μηχανισμός Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να γίνει αναφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, εκρίζωση της φτώχειας και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μακροπρόθεσμα ε, που αφορά την, ε, το χρονοδιάγραμμα για το 2030 θα πρέπει να διατυπωθεί σωστά ως βασικό πλαίσιο. Όπως πολλοί, ε, πολλοί από εσάς... Ε, τονίσατε το θέμα της ε, λογοδοσίας και της αξιολόγησης. Θεωρούμε ότι είναι αποδυναμωμένοι αυτοί οι μηχανισμοί. Θα πρέπει να υπάρχει μία αύξηση στην ευελιξία από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια δυσανάλογη, ένας δυσανάλογος εστιασμός της προσοχής στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να ακούσουμε και κάτι περισσότερο από τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχουν και ορισμένοι προβληματισμοί που αφορούν το θέμα της μετανάστευσης. Υπάρχουν θέματα που τα θεωρούμε απαράδεκτα και ελπίζουμε το ζήτημα της αιρεσιμότητας να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες που αφορούν τον κανονισμό και τα παρατήματα. Άφησα επίσης ε, αντίγραφα των τροπολογιών ε, για τα δικαιώματα των παιδιών. Βρίσκονται στο προστινό μέρος της αίθουσας και μπορείτε να τα πάρετε. Στην τροπολογία μας συμπεριλάβαμε μία σειρά από θετικά στοιχεία από τον υπάρχοντα κανονισμό που θα επιθυμούσαμε να διατηρηθεί. Για μερικά από αυτά ψηφίσατε εσείς. Υπάρχουν μερικές δικλείδες ασφαλείας που θα θέλαμε να επανεισαχθούν. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν πράγματα που υπήρχαν στο προηγούμενο κανονισμό και που έχουν ε, εξαφανιστεί. Ε, γιατί το ζητούμενο είναι ε, να έχουμε στο στόχο μας την ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεισαχθούν ορισμένα δεδομένα. Οι στόχοι ανάπτυξης δεν είναι επαρκείς και χρειαζόμαστε δικλίδες ασφαλείας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ο στόχος του 20% σε ό,τι αφορά τους γεωγραφικούς και θεματικούς πυλώνες και θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς θα ελέγχουμε αυτούς τους τομείς. Θα θέλαμε να ενδυναμωθούν αυτοί οι τομείς με βάση ε, τα άρθρα του κανονισμού. Υπάρχουν, ε, παρουσιάζουμε πάρα πολλές ε, ιδέες ε, στις τροπολογίες μας και στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το 20%. Το θέμα του φύλου μπαίνει κατά μέρο σε αυτή την προσέγγιση. Η ομάδα των γυναικών συμπιέζεται μαζί με την ομάδα των παιδιών. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι μοναδικές περιπτώσεις για επένδυση και νομίζουμε ότι θα πρέπει να αντικατοπρίζονται σε αυτό τον μηχανισμό. Δεν θα πρέπει να μνήονται αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο τομέων ε, δεν είναι προς όφελος της επίτευξης των στόχων μας. Εδώ μιλάμε για 20% δράσεις που απευθύνονται στο φύλλο. Οι, δύο, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να εσωματωθούν στον κανονισμό και να γίνουν σεβαστοί. Σε ό,τι αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι αρκετά επαρκής. Ας μην ξεχνάμε ότι μόλις τελείωσε ένα φοβερό καλοκαίρι με φοβερές ζημιές για το περιβάλλον. Τώρα ο στόχος είναι 50% και δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της ανάπτυξης που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω αυτού του μηχανισμού. Είμαστε η πέτσα, αναφορά στην κοινωνία των πολιτών. Παρόλα αυτά ο ρόλος κοινωνίας ε, των πολιτών δεν παρουσιάζεται επαρκώς σε αυτό το μηχανισμό. Θα θέλαμε να ε, εάν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν ενταχθεί στο γεωγραφικό πυλώνα, θα υπάρξει μια μεγάλη απώλεια κονδυλίων. Σε γενικές ε, γραμμές ε, παρατηρείται μια μείωση των κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά τον θεματικό πυλώνα, έχουμε μια έκθεση στην οποία ε, συγκρίνονται συγκρίσιμα στοιχεία και γίνεται μία αναφορά στις ε, παγκόσμιες προκλήσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης, η μετανάσταση ίσως ε, την χάνει δυσανάλογης προσοχής στο μηχανισμό. Η άποψή μας είναι ότι οι δράσεις θα πρέπει να έχουν μία μακρόπνοη προσέγγιση θα πρέπει να ενταχθούν σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να βοηθηθούν περιοχές που δέχονται μεταναστευτικές ε, πιέσεις. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες άμβλησης παράνομης ε, μετανάστευσης και ο, ο στόχος του 10% δεν αφορά μέτρα ε, που λαμβάνονται στα σύνορα έχουμε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει μία λανθασμένη χρήση αυτών των ε, μέσων. Και πραγματικά θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να έχουμε μία καρποφόρο συζήτηση για το μηχανισμό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ε, δύο συμμετέχουσες. Δίνω το λόγο στις, στους κοιόδους από τον Νόρμπερτ Νόιζερ. Ξεκινώ, μετά η κυρία Θεοχάρου, η κυρία Σαρτζεντίνη και η κυρία Σάντσε. κυρία Σοκοράου και ο, και ο Σαφχάουζερ. Ε, <clears throat> σας ευχαριστώ πολύ για τις σαφείς παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τους ε, εισηγητές μας και για το Κοινοβούλιο να παρουσιάζονται κάποια πράγματα με τέτοια σαφήνεια. Επικροτούμε την γεωγραφική προσέγγιση, επικροτούμε το ότι βρίσκονται στο επίκεντρο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα στην έκθεση, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να καθίσταται σαφής η θέση του Κοινοβουλίου ότι η απόλυτη προτεραιότητα έχει η καταπολέμηση της φτώχειας και ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, τις διατάξεις της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και θα πρέπει οι υπεύθυνοι ε, στις, χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες να φέρουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Όλα αυτά θα πρέπει να καθίστανται σαφή στην έκθεση. Communication pratique, euh, la cabine euh, portugaise est fermée pour cause de maladie. Ε, μια ε, ενημέρωση εξαιτία μια ασθένεια, η πορτογαλική καμπίνα διερμηνία θα κλείσει. Οπότε οι Πορτογαλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να ακούσουν ε, πορτογαλικά πλέον από εδώ και πέρα για σήμερα το πρωί. Εγώ θα συνεχίσω στα γερμανικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της καλής διακυβέρνησης, η ευθύνη της ελίτ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Επίσης θα πρέπει να περιγράψουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε στη μετανάστευση. Και εγώ πιστεύω ότι η μετανάστευση έχει να κάνει με όλα τα θέματα αυτά. Ως πολιτικοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη έχουμε βέβαια τη δική μας θέση πάνω στη μετανάστευση. Θα πρέπει να γίνουν πολλά για να ρυθμιστεί σωστά η μετανάστευση. Θα πρέπει όμως να ενεργούμε μακροπρόθεσμα και όχι απλά να λαμβάνουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναφερθήκατε στα δικαιώματα των παιδιών, ε, θέματα των δύο ε, την φόρο αποφυγή. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση και θα πρέπει να καθίσταται σαφές ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο νέο αυτό μέσο, το οποίο δίνει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, γενικά όμως είναι αρκετά ασαφές προς το παρόν. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Ο λόγος στην κυρία Σαρτζεντίνη. Η κυρία Θεοχάρους ε, απουσιάζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει συμπεριληφθεί εδώ, αλλά φαίνεται να μην έχουν συμπεριληφθεί τα σχετικά εχέγγυα. Κάποιος, κάποια από τις ομιλήτριες αναφέρθηκε σε αυτό. Μήπως μπορείτε να το αναπτύξετε αυτό. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο μέσο και αγωνιστήκαμε να υπάρχουν εχέγγυα ώστε να συμβάλλουμε στην εκρίζωση της φτώχειας. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς θεωρείτε ότι συμπεριλαμβάνεται αλλά παρά είναι γενικό. Ξέρω ότι είναι άποψη, αλλά θα ήθελα πολύ να την αναλύσετε. Επίση, όσον αφορά την παρουσίαση της κυρίας Ντόλμαν. Είπατε ότι ο ΣΑ έκανε πριν ε, κάποια χρόνια αξιολόγηση ομοτήμων και ότι κλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγχωνεύσει διάφορα ταμεία μεταξύ τους και να είναι πιο ευέλικτη. Δεν μα μιλήσατε όμως για το τι έχουμε μπροστά μας. Ναι, προφανώς έχουμε εδώ πέρα συγχώνευση, έχουμε και περισσότερη ευελιξία. Εγώ προσωπικά έχω αμφιβολίες σχετικά με το για ποιον είναι χρήσιμη αυτή η ευελιξία. Θα ήθελα όμως να μου πείτε γιατί κάνατε αυτή την έκκληση για συγχώνευση των ταμείων και περισσότερη ευελιξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάντσες. Ούτε η κυρία Σάντσες είναι εδώ. Ο κύριος Κορά επίσης, ο κύριος Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ευνηδιάζετε. Αλλά να σας πω μερικού προβληματισμού. μου. Καταρχήν πρέπει να στηρίξουμε την Αφρική. Αυτό αφορά ένα δισεκατομμύριο άτομα για το άμεσο μέλλον. Για αυτούς χρειάζεται να τους βοηθήσουμε να βρουν δουλειά, απασχόληση στις χώρες τους και αυτό απαιτεί, κατά την άποψή μου, μια ρύθμιση της οικονομίας και ένα βαθμό προστατευτισμού. Αυτό ισχύει και για μας, ισχύει και για αυτούς. Αν δείτε μάλιστα εμείς πώς αναπτυχθήκαμε στην ιστορία μας, πάντοτε είχαμε το δίλημα της ε, ανάπτυξης σε συνδυασμό με τον προστατευτισμό και του ελεγχόμενου ανοίγματο των συνόρων μας. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Δεύτερη σκέψη αφορά τα μέσα. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μέσα που χρειάζονται για να τροφοδοτήσουμε την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει μεταξύ του 2012 και του 2018 δύο δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε κρατικό χρέος σε διάφορα νομίσματα. δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και αυτό ισχύει και για τον Νότο, όπου, θα, όπου χρειάζεται οπωσδήποτε να επενδύσουμε για την δημιουργία καινούργιου πλούτου και όχι μόνο για τη λιτότητα, αλλά αυτό ισχύει και για την Αφρική. Τρίτη μου σκέψη αφορά τον τρόπο υλοποίησης των αναπτυξιακών μέτρων. Και αυτό ισχύει και για μας και για χώρες όπως η Αφρική. Ενιαία αγορά με νέο νόμισμα, ενισχύει τους πλούσιους και αδυνατίζει τους φτωχούς και τους αδύναμους. Θα έπρεπε λοιπόν, ειδικά για τις χώρες του Νότου, αλλά και για την Αφρική, να λάβουμε ιδιαίτερα μέτρα. Και στην Αφρική δεν παίζουμε με τα κράτη, αλλά πιο πολύ με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που όμως ποτέ δεν θα γίνουν φορείς ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε πώς οργανώνουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε κύριε Σαφχάουζερ. Ο λόγος τώρα στους ευρωβουλευτές, η κυρία Λόζινγκ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω ότι πολλοί από αυτούς ε, τους στόχους καθορίζονται από κοινού από όλους μας ε, με συνένεση. Μιλάμε εδώ για διάφορες πτυχές της χρηματοδότησης. Ε, γι' αυτό θα προσπαθήσω να εστιάσω ακριβώς στις πτυχές αυτές. Θα ήταν θετικό αν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πάντα μιλάμε για την ευελιξία. Συνάδελφος από την Επιτροπή Ανάπτυξης έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για ευελιξία και τι επιπτώσεις πρακτικές μπορεί να έχει αυτό. Είμαι μέλος της ΑΦΕΤ. Και από αυτήν την οπτική βλέπω το θέμα της συγχώνευσης των διαφόρων ε, ε, μέσων της εξωτερικής πολιτικής. Και σκέφτομαι ιδιαίτερα την συγχώνευση της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της ε, πολιτικής άμυνας. συνάδελφος του S&D αναφέρθηκε και στη μεταναστευτική πολιτική. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι πόσο χρήσιμο είναι για μια βιώσιμη πολιτική ανάπτυξης η καταπολέμηση της μετανάστευσης Κατά πόσο δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε στην μεταναστευτική πολιτική, διότι αν εξετάσουμε τα επιμέρους μέσα, διαπιστώνουμε ότι όλο, και περισσότερα χρήματα για την ε, καλή διακυβέρνηση ή για την ανάπτυξη ε, δαπανώνται τελικά για την ε, προστασία των συνόρων, για την συνεργασία με, τα, με τις χώρες της Αφρικής με τον στόχο του περιορισμού της μετανάστευσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν στο NDICI πόσο χρήσιμη είναι αυτή η συνεργασία και κατά πόσο έχει στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα ήθελα να ακούσω κατά τη γνώμη σας η συγχώνευση της πολιτικής ασφάλειας κάθετος πολιτικής μετανάστευσης θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας. Και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί με την συγχώνευση αυτή που γίνεται με σλόγγαν την ευελιξία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ θερμή παρέκκληση να γίνεται σεβαστός ο χρόνος αγόρευσης των δύο λεπτών. Χάιντι Οτάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε λόγο να προβληματιζόμαστε ότι θα προκύψουν μερικά ωφέλη, δηλαδή θα μπορούσε να καλεί αυτή η ευελιξία. Πραγματικά πιστεύω ότι το να προσεγγίσει το γεωγραφικό, το θεματικό πρόγραμμα είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να καούν τα, χλωρά μαζί με τα ξερά. Η εκρίζωση της φτώχειας δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να <clears throat> προωθήσουμε αυτή την άποψη. Έχω μερικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά το μηχανισμό που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ειρήνη, ο οποίος βρίσκεται εδώ μέσα. Με εκπλήσει το γεγονός ότι μία σειρά από στόχους και δράσεις δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στον κοινό μηχανισμό. σχεδόν 22 πολιτικές έχουν διαγραφεί και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των ειδικών. Ποιος θα πρέπει να είναι στόχος ε, αυτού του μηχανισμού σε ό,τι αφορά τη συμβολή του στη σταθερότητα και στην ειρήνη. Για ποιο λόγο γίνεται εστιασμός της προσοχής στην αύξηση των στρατιωτικών ικανοτήτων. Εμένα με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα πρόταση ε, για ένα μηχανισμό ειρήνη, ειρηνευτικό μηχανισμό και δεν θέλω να γνωρίζω ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών για σας. Τέλος ακούσαμε να γίνεται αναφορά σε μια σειρά από σημαντικές αρχές του ΟΣΑ για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά την άποψή σας υπάρχουν στοιχεία αυτού σε αυτό το μηχανισμό. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτό το μηχανισμό. Δηλαδή πόσο καταφέρει να εφαρμόσει τις αρχές που εσείς προαγάγετε. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, η κυρία Λίντα σε ευχαριστώ, Σάρλιν. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για την Επιτροπή και όχι για τους προσκεκλημένους ομιλητές. Θα πάρει το λόγο μετά η Επιτροπή. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι, με το ότι αυτό που λείπει είναι ο τονισμός των στόχων στην, ε, στο γενικό χρονοδιάγραμμα. Και αναρωτιέμαι αν η Επιτροπή θα μπορούσε να μας πει τι συμβαίνει. Συνδυάζουν πολλούς μηχανισμούς. Κατά την άποψή τους υπάρχει κάτι αρνητικό στο να ενδυναμωθεί αυτή η πτυχή είναι η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τα Κορίτσια και η Επιτροπή είπε ότι θα έχουμε να κάνουμε με τον πιο α, φεμινιστή ε, επίτροπο. Σύμφωνα με όσα συμφωνήσαμε ε, στο παρελθόν, τι συμβαίνει εδώ. Σε ό,τι αφορά τις κλιματικές ε, αλλαγές, ακούσαμε την έκθεση IPCC και νομίζω ότι είναι σαφές από αυτή την έκθεση ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα. Ε, έχω ένα ερώτημα για τον ΩΣΑ τώρα, αλλά και για την Επιτροπή. Είναι εύκολο να λέμε για την εξωτερική πολιτική ότι θα πρέπει να είναι, παρουσιάζει συνοχή. Αλλά οι εγχώριες πολιτικές, οι εσωτερικές πολιτικές, ε, πόση συνοχή έχουν με από μερικά χρόνια. Υπήρχε ένα λόμπι που έλεγε ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εργοστάσια άνθρακα στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες λόγω της ε, ε, Εδώ όμως χρηματοδοτούμε τα καύσιμα. Μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια, να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε και μια συνοχή. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στο εσωτερικό κάνουμε ό,τι και στο εξωτερικό. Δηλαδή στην ουσία να μην είμαστε δάσκαλοι που δίδασκες. Μήπως η Επιτροπή θα μπορούσε να μας πει ε, τι θα κάνει, αν θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο, αν θα διαπραγματευτεί για τις εκπομπές των αυτοκινήτων. Αν θέλουμε να στείλουμε ένα σωστό μήνυμα, θα πρέπει και μεταξύ μας να έχουμε συνοχή και συνέπεια. Θα ήθελα η Επιτροπή να μου μιλήσει για τα κονδύλια για τα CFOs. Ξέρω ότι θα μου τεθεί ερώτηση για το CSO, ε, φαίνεται ότι έχει μειωθεί. Η Επιτροπή μετά όμως ε, μου λέει από την γεωγραφικό, το γεωγραφικό ε, σκέλος θα υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διευκρίνηση από την Επιτροπή και για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά το FSD, Νομίζω ότι είναι ένα μέσο, ένας μηχανισμός που θα ενταχθεί τώρα στο καινούριο πρόγραμμα. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε από άποψη επενδύσεων, τι θα αλλάξει, τι θέλετε να αλλάξετε, τι θέλετε να έχετε στο μέλλον υπάρχουν ομάδες πίεσης, αλλά εσείς πέστε μου τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το επενδυτικό τοπίο. Ε, ήμουν στην Γκάνα την ε, ε, προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να να δουν περισσότερες επενδύσεις, όχι μόνο απλές ενισχύσεις. Θα ήθελα να ε, αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Τι πρακτικό λοιπόν γίνεται εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λίντα. Στου συνάδελφου Πρέντα, συνεισηγητήσα. Ευχαριστώ Σάλ. Ως μέλος της Επιτροπής ΔΕΒΕ θα πάρω το λόγο αν μου επιτρέπεις. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση πολιτικής φύσεως η σημασία της Αφρικής υπογραμμίστηκε. Η συνοχή των πολιτικών μας για την Αφρική επίσης. Θέλω να πω το εξή όμως. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην Αφρική, αλλά δεν θα πρέπει να θυσιάσουμε ένα κομμάτι της πολιτικής γειτονίας, αυτό που αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει ο πειρασμός. Οι γειτονικέ χώρες του Νότου να μετατραπούν σε κάποιους, σε χώρες που νεοαφιχθήσεις στην Αφρική. Αυτή είναι μια λάθος κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να δώσουν περισσότερο ρόλο στην Αφρική σβήνοντας τις σχέσεις μας με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την καρεβική και τον Ειρηνικό, τις χώρες ΑΚΕ, το υπόλοιπο των χωρών ΑΚΕ δηλαδή. Στην πολιτική μας, ε, στο παρελθόν, είχαμε βάλει στην ίδια ομάδα όλες αυτές τις χώρες, χώρες ΑΚΕ. Δεν θα πρέπει η ιδιαίτερη σημασία που θα δώσουμε στην Αφρική να μας οδηγήσει στο να ξεχάσουμε την Καραβική και τον Ειρηνικό. δεν θα πρέπει οι προτάσεις για τον καινούριο μηχανισμό να αλλάξουν τις ισορροπίε που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Βέρκα Πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να αυξηθούν τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κονδύλια για την ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φτώχειας στην Αφρική. Και είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εμπορικές συνεργασίες. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το μέρος της πρότασης. χρηματοδότηση της ε, ανάπτυξης ε, θα μπορούσε να έχει ως σημείο εκκίνησης ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας και της συνεργασίας. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι πολλά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν την ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Δημερός. Τι είδου συντονισμός γίνεται σε ό,τι αφορά την εθνική χρηματοδότηση. Όταν δίνουμε χρήματα από τα ενωσιακά κονδύλια, από τη μία πλευρά υπάρχουν τα ενωσιακά κονδύλια και οι χώρε μέλη δοτούν ξεχωριστά. Τι είδου συντονισμό γίνεται σε ό,τι αφορά την εθνική και ενωσιακή συνεργα... Ε, χρηματοδότηση, κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσοι εισηγήτρια για την νομοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η κυρία Άλβα Φίν εξ ονόματος της Κόγκον σχετικά με διάφορα σημεία. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν οι υπόψη η νοικιό και η κοινωνία των πολιτών ως συνομιλητές. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν μακρόπνοες πολιτικές που επιδιώκουν την εκρίζωση της στόχιας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των κλιματικών καταστροφών. Συμφωνώ με τα ερωτήματα που ετέθησαν σε ό,τι αφορά το θέμα της ευελιξίας. Αυτό που θα ήθελα να αποφευχθεί είναι το να μην δώσουμε, να μην ανταποκριθούμε στις πιο πιεστικές ανάγκες των πιο ευάλωτων χωρών, ας πούμε Νότιο Σαχάρα και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Φοβάμαι ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε στόχους εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι ο στόχος ε, θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και όχι στρατηγικές επιλογές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι κατά ε, του συσχετισμού της αιρεσιμότητας ανάπτυξης με την άμυνα και τον έλεγχο της μετανάστευσης. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την πρόταση της Επιτροπής ε, που αναφέρεται στη σκοπιμότητα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν λαμβάνονται αποφάσεις ε, κυρίως ε, έκτακτου χαρακτήρα, όταν δίνονται έκτακτες ενισχύσεις. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να αποκτήσει τη δυνατότητα να ελέγχει ε, Τέλος, πιστεύω ότι για τους λόγους που προανέφερα θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του θεματικού πυλώνα και του γεωγραφικού πυλώνα. Ο γεωγραφικός πυλώνας εξαρτάται περισσότερο από γεωπολιτικές επιλογές που είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά όχι κατά ανάγκη των πιο ευάλωτων χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον οποίο αναφερθήκατε ε, είναι πολύ σημαντικός. Αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να υπερασπιστούμε αυτό το ρόλο. Η τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Σόλτ. Ενάμιση λεπτό σας παρακαλώ. Γιατί δεν θα υπάρχει χρόνος για να δοθούν απαντήσεις. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο απόψεις θα ήθελα να εκφράσω. Αναφέρθηκε η ευελιξία και το mainstreaming, η απλούστευση. Η κυρία Φιν πολύ σωστά είπε ότι η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς μας και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς με όλα αυτά τα μέσα καταφέρουμε τον στόχο μας όταν ε, ε, δεν υπάρχει συνεκτικότητα ανάμεσα στα ε, διάφορα μέσα. 1,3% είναι το ποσοστό της χρηματοδότησης και παραμένει το mainstreaming το βασικό κριτήριο για την βιώσιμη ανάπτυξη και έχουμε περιορισμένο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των στόχων αυτών. και δεν θα πρέπει απλά να ασκούμε πολιτική ανάπτυξη για άλλους. Θα πρέπει να, να αλλάξουμε ε, τα ε, πρότυπά μας ώστε το 2050 οι άνθρωποι στην Αφρική να ε, έχουν τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσης. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι σταγόνες στον ωκεανό. Και η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε έλεγχο των μέσων, έλεγχο των πόρων στα μέσα αυτά. Και μάλιστα οι επιτροπές ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε διορθώσεις στην κατανομή των μέσων και γι' αυτό είμαι κατά της έκδοσης κατεξοδότηση πράξεων θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να τα κάνει αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές από, καταρχήν από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι δύσκολο να απαντήσω σε όσα, σε ελέγχθησαν και να δώσω και, και απαντήσεις στα σχόλια. Και... πάση περιπτώσει όμως θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την ακρόαση. Είναι πολύ χρήσιμο. Όπως και εμείς είμαστε εδώ από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και έτσι και εσείς ε, οι δύο επιτροπείς ε, ε, ΑΦΚΟ και ΕΝΤΕΔΕ, είσαστε μαζί και αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης είναι εξαιρετική ιδέα αυτά τα δύο πάνελ, γιατί στην πραγματικότητα προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ίδιο ερώτημα, πώς θα παραμείνουμε παγκόσμιος παίκτη, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την επιρροή που έχουμε στην παγκόσμια σκηνή, διατηρώντας τις αξίες μας, σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση, τους κανόνες και το έργο μας. Και όλα αυτά προσπαθούμε ήδη να τα απαντήσουμε με την μεταρρύθμιση του μηχανισμού. Η απάντηση όμως στην πραγματικότητα είναι η Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 δεν αφορά πλέον μόνο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή 15 κρατημέλη μιλούν. Για παράδειγμα Γερμανία, Φιλανδία, Ισπανία, Παρίσι και Χάγη. Ε, έχουμε 15 χώρες οι οποίες ασχολούνται πολύ εντατικά με την Ατζέντα 2030, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις χώρες στις γειτονικές μας και τις πιο μακρινές, τη Λατινική Αμερική κλπ. Οπότε η Ατζέντα αυτή έχει πάει πολύ μακριά. Τη στήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δική σας συνεργασία και με τη συνεργασία των ομιλητών σήμερα. Προσπαθούμε να την προασπίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Συνεργαζόμαστε λοιπόν πλέον με τα κράτη-μέλη αλλά και με τον ΟΗΕ για να προωθήσουμε κοινό προγραμματισμό προκειμένου να βοηθήσουμε τις τρίτες χώρες να εισάγουν στη δική τους πολιτική την Ατζάντα 2030 με δείκτες, με πολιτικές, με στόχους. Και μια πολύ καλή εισαγωγή είναι ε, ότι αυτό θα πρέπει να μπει και στην εξωτερική μας πολιτική. Αλλά και εσωτερικά. Ε, για παράδειγμα, γεωρική πολιτική και η συνοχή των πολιτικών μας, ο ε, κρόσπι θα διανοηθεί την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να το δούμε και με τα κράτη-μέλη. Εσωτερική λοιπόν συνοχή των πολιτικών μας, διότι δεν πρέπει εμείς απλώς να το ζητούμε, αλλά θα πρέπει να γίνει πράξη όλες οι εσωτερικές πολιτικές, εμπορική πολιτική, εμπορική πολιτική κλπ. να ειδωθούν από την πλευρά της συνεκτικότητάς τους. Τρίτον, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που είπαν, νομίζω πως η πρόταση της Κομισιόν για το μηχανισμό γειτονία ανάπτυξη και διεθνούς συνεργασίας έχει κάποια προβλήματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά είναι καλή πρόταση, είναι καλή βάση εργασία, διότι περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία και αντιμετωπίζει τη δράση μας με ένα πιο ευρύ και σφαιρικό τρόπο. Μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, φύλλο, όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το μηχανισμό. Άκουσα κάποια σχόλια για το κατά πόσον η Ατζέντα 2030, το φύλλο, η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικόματα κλπ. κλπ. μπορούν να τονιστούν περισσότερο. Όλα αυτά μπορούν ασφαλώ να γίνουν, θα τα εξετάσουμε μαζί. Θα ήθελα να ρωτήσω του εμπειρογνώμονε, ξέρετε αν υπάρχει κάποιο κράτο μέλο που ε, μέσω του νόμου έχει θέσει το στόχο του 85% για ε, για τις δράσεις ε, τις σχετικές με το φύλλο ή κάποιο άλλο στόχο ο οποίος να έχει ε, εδρεωθεί μέσω ενός νόμου. Εμείς ως Κομισιόν θα στηρίξουμε τους στόχους σε σχέση με το φύλλο κλπ. Αλλά δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά κανένα κράτος μέλος που να έχει εισάγει στην ομοθεσία τέτοιου είδους κανόνες, τέτοιου είδους ποσοστά και στόχους. Κάποια άλλα πράγματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το EFSD. Το καινούριο EFSD ε, έχει καινούριους κανόνες. Το μελλοντικό EFSD θα έχει 92% των πόρων του τα οποία θα δίδονται με βάση ε, κανόνες λογοδοσίας. Αυτή τη στιγμή υπόκειται σε όλους τους κανόνες που έχουμε ε, και για το μηχανισμό ε, χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Έχουμε όλους τους ίδιους κανόνες και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Τώρα πλέον ισχύουν και αυτοί οι κανόνες. Δεν είναι λοιπόν εξαίρεση το ΙΕΦΕΣΤΗ. Για ποιο λόγο? Γιατί αντίθετα με τη σημερινή κατάσταση οποιοδήποτε τέτοιου τύπου ταμείο δεν θα χρηματοδοτεί εξ αρχής δράσεις ε, οριζόντια, αλλά με βάση γεωγραφικά προγράμματα, τα οποία θα διέπονται από συγκεκριμένες προτεραιότητες, τις οποίες θα ορίσουμε σε συνεργασία με τις χώρες που είναι οι δικαιούχοι χώρες. Τέλος μετανάστευση και ασφάλεια. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη μετανάστευση στην Κένια, αλλά όχι, ε, αλλά λέτε εσείς, αλλά μπορούμε να δούμε τη μετανάστευση στο Περού για παράδειγμα. Γιατί, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η Κένια. Δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά. Έχετε δει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το καταπιστευματικό ταμείο και νομίζω ότι το κάνουμε καλά. Τέλος, για τις γεωγραφικές και θεματικές επιλογές. Ναι, βάζουμε περισσότερη, ε, δίνουμε περισσότερη σημασία τη γεωγραφική κατανομή γιατί θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Μας βοηθάει αυτό επίσης να συντονιστούμε καλύτερα με τα κράτη-μέλη και να εφαρμόσουμε την Ατζέντα 2030 αναχώρα καλύτερα. Έτσι θα ακούσουμε καλύτερα και τις χώρες που είναι δικαιούχες. Η, η θεματική κατανομή διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όχι τις δικαιούχες χώρες. Αυτά για από μένα Έχω και κάποιους συναδέλφους που θα ήθελαν το λόγο να απαντήσουν σε κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία τέθησαν στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πολύ λυπάμαι ότι θα χρειαστεί να διακόψω τους επόμενους ομιλητές ε, γιατί ο χρόνος ε, πιέζει πάρα πολύ και έχουμε και ένα δεύτερο πάνελ. Ο κύριος Φίλιπ Μπερτό Σεριάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχάς, θερμές ευχαριστίες και οι δύο παρουσιάσεις ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και πραγματικά Ειδικά μου άρεσε το ότι εστιάστηκε η ε, προσοχή προς τις θετικές εξελίξεις και υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και των μηχανισμών. Ένα σχολισμό, σχολιασμός για την ε, ε, συνοχή των πολιτικών. Έγιναν ορισμένα σχόλια για την εμπορική πολιτική, για την γεωργική πολιτική, για το τι θα συμβαίνει αυτό από την άποψη ενός συμβιβασμού. Θα ήθελα να πω κάτι που συχνά λέει και η ύπατη εκπρόσωπος Μοργέινη. Όταν τίθενται θέματα όπως ασφάλεια και μετανάστευση, ο φόβος μας είναι ότι αυτές οι πολιτικές και θα μπορούσαν να απορροφήσουν κονδύλια από την ανάπτυξη. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το δούμε το θέμα και από την αντίθετη οπτική γωνία. Αν δούμε τι κάνουμε για να στηρίξουμε το, ε, την Αφρική, το Σαχέλ, αυτό σημαίνει ότι στην ουσία αυτό που θεωρείται ως θέμα μετανάστευσης ή ασφάλειας έχει σχέση με την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης και της έλλειψης σταθερότητας. Δηλαδή στην ουσία εστιάζεται προς την στήριξη της ανάπτυξης και της ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε με έναν θετικό και όχι με έναν αρνητικό τρόπο. Δεύτερον, εκφράστηκαν κάποιοι προβληματισμοί όσο προς το κίνδυνο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε βραχυχρόνιες και όχι μακροχρόνιες προοπτικές. Το 75% των πόρων θα πάνε σε γεωγραφικά προγράμματα και αυτό θα είναι το πρόγραμμα μακροπρόθεσμα, δηλαδή θα ε, ασχοληθούν με μακροπρόθεσμα ε, θέματα και ο προγραμματισμός θα είναι μακροπρόθεσμος. Και όπως είπαμε, τον 92% κατά την άποψή μου βρίσκεται για να μας δώσει διαβεβαιώσεις σε ό,τι αφορά το μακροχρόνιο με το βραχυχρόνιο. Από την άλλη ε, πλευρά το να υπάρχει ένας ενδιάμεσος πόρος, οι πόροι που μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες ε, καταστάσεις ε, δεν μπορεί να είναι παραθετικό σε ό,τι αφορά την ικανότητα δράσης μας στο, ε, γενική, στην ε, ε, παγκόσμια σκηνή. Επίσης με ικανοποίησαν μερικά σχόλια σχετικά με το συνδυασμό των δράσεων των χωρών μελών. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν κοινά προγράμματα και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Το τελευταίο σημείο αφορά την αναφορά που κάνατε στην ανάγκη για τακτική ενημέρωση και έλεγχο από πλευράς του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το νέο αυτό μηχανισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία πιο τακτική ανταλλαγή πληροφοριών που ε, συνδέεται με θέματα πολιτικά και όχι με θέματα διοικητικά τόσο πολύ και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές για το Κοινοβούλιο. Τέλος, έγινε μία αναφορά σε στόχους της πολιτικής, τους οποίους δεν επιτυγχάνουμε. Ο, η βάση εδώ είναι ότι οι πολιτικές ορίζονται στα έγγραφα και ε, το, ενώ το άλλο είναι ένα οικονομικό εργαλείο. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί βεβαίω με βάση τις δικές σας υποδείξεις. Η μοναδική μου προειδοποίηση, ας αποφύγουμε να έχουμε ένα υπερβολικά υψηλό αριθμό συγκεκριμένων στόχων, διαφορετικά ένας ενιαίος μηχανισμός ε, θα παγιδευτεί μέσα σε αυτό το πλέγμα των δίσκαμπτων στόχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο λόγος στον κύριο Χάντς Γιάνσεν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο εδώ όπως είπατε. Ε, λέγομαι Hans Janssen. Ε, έρχομαι από μια περιοχή κοντά στο Eindhoven στις κάτω χώρες και θα ήθελα να απαντήσω εδώ στις σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις ε, προτάσεις που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή. Πρόκειται για σημαντικές και φιλόδοξες προτάσεις. η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ε, η ε, εκρίζωση της φτώχειας, ε, η μετανάστευση είναι σημαντικές προκλήσεις. Έχει τονιστεί ο ρόλος των τοπικών αρχών, κάτι που επικροτούμε. Έχουμε όμως και κάποιες ανησυχίες. Για παράδειγμα, δεν βλέπουμε να αναφέρεται ο, ο προϋπολογισμός για τις ε, τοπικές αρχές. Αναφέρονται, δεν αναφέρεται όμως η δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω γιατί έχει γίνει αυτό. Ε, εάν δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση των ε, πόρων αυτών, αυτό μπορεί να οφείλεται με τις υψηλές απαιτήσει για την συγχρηματοδότηση. Για να πετύχουμε θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση. Το μεγάλο δεν είναι πάντα ωραίο. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Και έτσι φτάνουμε στον πυρήνα της συζήτησης για την ευελιξία. Κύριε Πρόεδρε, οι έρευνες έχουν δείξει ότι το 25% των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί ε, με την εμπλοκή των τοπικών αρχών που βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Η έκκληση μου λοιπόν είναι όταν μιλάμε για πολιτική γειτονία ή προενταξιακή πολιτική, οι ευρωπαϊκοί κανόνες θα πρέπει να επιτρέπουν και την συμμετοχή των ε, αρχών στο πιο χαμηλό επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη των ε, στόχων του 2030. Ελπίζω να μπορέσετε να υιοθετήσετε την πρότασή μας ε, και να ασκήσετε κι εσείς πίεση. Κυρία Ναντίν Κρίσεστεν, εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Έχουμε να κάνουμε τα παρακάτω σχόλια και συστάσεις. Όπως είπαν πολλοί από τις προηγούμενες ομιλητές, εμείς θα συστήναμε σε ό,τι αφορά την, τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης να τονιστούν περαιτέρω σε όλο τον κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη την αρχή του να μην μένει κανείς πίσω. Μια αρχή βαθιά ριζωμένη στην Ατζέντα 2030. Επίσης θα συστήναμε ε, να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του πιο ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού ανεξάρτητα από το που ζουν. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα και θα θέλαμε να πούμε ότι το 75% δίνουν προτεραιότητα στο γεωγραφικό πυλώνα, μόνο 8% το θεματικό πυλώνα. Ο δικός μας προβληματισμός είναι ότι αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγγυήσει ότι τομεί που συμπεριλαμβάνονται στο θεματικό πρόγραμμα όπως υγεία, ανάπτυξη, δεξιότητες θα αποκτήσουν προτεραιότητα στο γεωγραφικό πυλώνα από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επιθυμούσαμε να συνεργαστούμε έτσι, για, να έχουμε την βεβαιότητα ότι αυτό θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό και το μηχανισμό. Σε ό,τι αφορά το 20% για κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη, βλέπουμε ότι το σχέδιο, στο σχέδιο κανονισμού αναφέρεται στο κοινωνικό, ε, στην κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ πιο ευρύ στόχο σε σύγκριση με το 20% στο ε, του EDCI. Εμείς είμαστε υπέρ του να διατηρηθεί ένα 20% για την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και να υπάρχει μια μεθοδολογία μέτρησης του σημείου αναφοράς. Θα συστήναμε την ανα... το να υπάρξει ένα σωστό ορισμό ε, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης με σαφή αναφορά στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία. Κοιτάζοντας το θέμα του φύλου, θα ήθελα να πω ότι ότι γίνεται αναφορά στο θέμα της ισότητας ε, ε, των φύλων και της αντινάμωσης των γυναικών, θα θέλαμε να συστήσουμε μία πιο άμεση προσέγγιση μέσα στη σύσταση, αλλά και να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα σημεία αναφοράς που έχουν σχέση με την ισότητα και σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης και η ισότητα μεταξύ των δύο πύλων να συμπεριληφθεί στους συγκεκριμένους στόχους του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, τα Ηνωμένα Έθνη στις Βρυξέλλες θα ήθελα να τονίσουν τη σημασία που έχει η άμεση επένδυση στους περιβαλλοντικούς στόχους και ε, ε, το θέμα της προσαρμογής στο κλίμα. Ε, τέλος, θα λέγαμε η οικονομική ενίσχυση που δίνεται στο κανονισμό να στηρίζεται ε, ε, στον στόχο της ε, ε, του αντιμετώπισης του θέματος της μετανάστευσης και των πρόσφυγων. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στα δύο άτομα τα οποία μίλησαν καταρχήν ε, σε αυτό το πάνελ, την κυρία Ντόλμαν και την κυρία Φιν. Κυρία Ντόλμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έγινε μια ερώτηση για τον ΟΣΑ και τις συστάσεις του του 2012 και τις πιο πρόσφατες. Η οπτική του ΟΣΑ για αυτό το θέμα θα είναι αποτέλεσμα μιας ευρεία συζήτησης μεταξύ των δωρητρίων χωρών του ΟΣΑ. Αυτή η άποψη θα υιοθετηθεί μετά την 24η Οκτωβρίου που θα γίνει η συνάντηση ε, αξιολόγησης. Για το θέμα που έθεσε η Λίντα Μακάβαν και άλλοι για την σημασία λήψης εσωτερικών μέτρων συνοχής πολιτικής, πολιτικών. Πάντοτε υπήρχε αυτή η ανάγκη. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη εν μέρη εξαιτία της θεσμικής δομής. Οι συντονιστές τη συνοχή των πολιτικών πολύ συχνά εργάζονται στο, στα Υπουργεία Εξωτερικών και σε εθνικό επίπεδο είναι δύσκολο αυτοί να βάλουν σε τάξη τους εκπροσώπους των υπολείπων Υπουργείων από την αρχή της ε, διαμόρφωσης της πολιτικής πρέπει η συνοχή των πολιτικών να ενταχθεί στην διαδικασία λήψη αποφάσεων από τα πρώτα στάδια. Ευχαριστώ. Um, for ε, κυρία Φιν, ευχαριστώ πολύ για την στήριξη που λάβαμε ε, ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στο φύλλο, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Ε, για την ευελιξία, όλα αυτά έχουν σχέση με την ευελιξία. Ένας ευρωβουλευτής είπε ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να συνδεθούν αυτά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ασφαλώς, ακόμα και οι μηχανισμοί ε, ευελιξίας θα πρέπει να έχουν μια λογοδοσία ένα κομμάτι λογοδοσίας. Ίσως η Κομισιόν δεν κατάλαβε πολύ καλά ποια ήταν η άποψή μα για το γεωγραφικό έναντι του ε, θεματικού. Ε, δεν θα πρέπει να το ένα να λειτουργήσει βάρος του άλλου, θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Η μείωση της θεματικής προσέγγισης έχει σχέση με την βελτίωση της ευελιξίας. Συμφωνούμε με την γεωγραφική προσέγγιση, όμως χρειάζεται ίσως λίγο λιγότερη ευελιξία έτσι ώστε ο θεματικός πυλώνας να γίνει πιο χρήσιμος. Γιατί αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση είναι πολύ μικρή πια για αυτό τον πυλώνα. Ετέθησαν κάποια θέματα σε σχέση με το πώς θεωρούμε ότι θα να ενισχυθεί η εκκριζωστή στόχια, η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. Έχουμε κάνει κάποιε τροπολογίε για το άρθρο 3. Στόχοι και επίση στο, στο άρθρο 8 για τι αρχέ. Αυτές οι τροπολογίες αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα κατά πολέμηση των ενισοτήτων, της φτώχειας, ε, ε, έμφαση στις ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Κάποιος είπε ότι οι μη κυβερνητικέ δεν θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Ε, εγώ θα σας πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η δική μας, το Save the Children, ε, λειτουργούν εδώ και 100 χρόνια, έχουν τεχνογνωσία την οποία δεν έχει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι κυβερνητικέ οργανώσει και η κοινωνία των πολιτών είναι κλειδιά προκειμένου να διαμορφωθούν πολυφωνικές δημοκρατικές κοινωνίες. Οπότε πιστεύουμε ότι ο ρόλος του θα πρέπει να ενταθεί, να ενισχυθεί. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο σχολιάσε η Κομισιόν, από το εξή. Ο κανονισμός του EFSD αναφέρει τη λογοδοσία. Και εκεί αναφερόταν ήδη ότι θα πρέπει, θα έπρεπε όλες οι δράσεις να τηρούν τους κανόνες του όσα Αυτό θέλουμε να επαναληφθεί στον καινούργιο κανονισμό. Επίσης, το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να ειδωθεί από την πλευρά της ανθρώπινης ασφάλειας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και όχι ως άμυνα ενός κράτους. Γιατί αλλιώς θα μειωθεί το στοιχείο της ανάπτυξης. Τέλος, το κατά πόσον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν μέσω των κάποιων στόχων βιώσιμης, στόχων ανάπτυξης για ε, την έμφαση σε θέματα όπως του φύλου κλπ. Η Αυστρία το έχει στο σύνταγμά της. Ο λόγο για τον οποίο δεν πετυχάνουν οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη είναι ακριβώ επειδή δεν έχουν ενταχθεί σε ένα νόμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή. Είδατε τι έγινε χτε ε, με τι αποκαλύψει και, ε, και την έρευνα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Φρανκ μπορεί να σας αναφέρει τα συμπέρασματα τα οποία βγάζει, είναι και Λουξεμβούριο. ξέρει να συμβιβάζει τις καταστάσεις. Ε, δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Αγγέλ. Κυρίες, κυρίες ε, και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, μόλις επέστρεψα από μία επιτροπή, ε, από μία αποστολή, με συγχωρείτε. Σημείωσα τρία σημεία που θα επιθυμούσα να θίξω στην τελική αυτή παρέμβαση. Θέματα που, στα οποία αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παρεμβάσεις. Μετανάστευση. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αναγκαστικά θα υπάρχουν βαθύτερες επιπτώσεις στο μέλλον, μια βαθύτερη εμπλοκή στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την διαχείριση του παγκόσμιου μεταναστευτικού φαινομένου, αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε σε μια παγκόσμια ε, αντίληψη και αυτό θα εμπνεύσει αρκετές από τις πολιτικές μας αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε τομεακές πολιτικές που δεν έχουν καμία σχέση με τη μετανάστευση ή να κάνουμε σαν να μην έχει καμία σχέση μετανάστευση με άλλες πολιτικές που υιοθετούμε. Ο συγκεκριμένοι στόχοι είναι το άλλο θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να ελέγξουμε αν συνεχίζουν πολλά ε, να, ισχύουν, να ισχύουν πολλά από τα πιστεύω μας. Δεν μπορούμε να ε, εκριζώσουμε τη φτώχεια έτσι, μοιράζοντας καρτονομίσματα. Εάν δεν λειτουργεί το κράτος, ε, δεν μπορεί να εκριζωθεί η φτώχεια. Δεν εκριζώνεται η φτώχεια αν δεν προσεγγίζουμε τον πληθυσμό που θέλουμε να βοηθήσουμε εκεί όπου ζουν, εκεί που ε, ε, ε, γίνονται μάρτιες σε ένοπλες σειράξεις. Θα πρέπει άλλα να μας εμπλεύσουν για το, την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Ας δούμε τον Νίγηρα. Ο Νίγηρας από τον Ήγηρα το 6% των συναλλαγών περνάνε από τις τράπεζες. Οι υπόλοιπες ε, συναλλαγές γίνονται όσα. Αυτό σημαίνει ότι το 94% των εμπορικών ε, συναλλαγών δεν υφίστανται κανέναν έλεγχο, καμία φορολογία. Δεν μπορεί να γίνει καμία ανακατονομή. Πώς εγώ θέλω να κρυζώσω την ε, ε, φτώχεια σε μια χώρα που έχει δημοκρατική, ε, ανάπτυξη 4%. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε, όπως φαίνεται το θέλει και η Επιτροπή, ότι η μία ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της πολιτικής ανάπτυξης. Δύο λόγια για τη γεωγραφική προσέγγιση. χιλιάδες φορές ε, είπαμε ότι χρειάζεται μια στρατηγική με την Αφρική, για την Αφρική. Χρειάζεται μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης Αφρικανικών Κρατών. Τώρα οι πολιτικές που εφαρμόζουμε δεν γνωρίζουν την ε, διάσταση της Αφρικής και προσπαθούν να τη δημιουργήσουν προσπαθώντας ε, ε, να συγκεντρώσουν κονδύλια για να μπορέσουν να, αντιμετωπίσουν την Αφρικανική Ήπειρο στο σύνολό της. Καταβάλλοντας παράλληλα μία προσπάθεια να ε, διατηρηθεί η παρούσα σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Γιατί κανένας δεν είπε ότι η λογική το χωρών ΑΚΕ θα πρέπει να εξαφανιστεί εντελώς αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την Αφρική στο σύνολό της, νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ότι η Καραϊβική ανήκει στην Αμερική, ο Ειρηνικός ανήκει στην ε, Ασία. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ ε, έχουν ε, γίνει επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές της Κόρης και, και αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να έχουμε κατά νου στην έκθεση. Μίλησα 24 δευτερόλεπτα παραπάνω από το χρόνο αγόρευσης που μου είχε δοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας ε, σε αυτό το πρώτο πάνελ και να ευχαριστήσουμε και τους συνεισηγητές μας. Θα αλλάξουμε πάνελ τώρα για το δεύτερο ε, μέρος ε, της ακρόασης. Έχουμε καθυστερήσει, συνάδελφοι, και έχουμε χρόνο μέχρι τις 11.30 ακριβώς. on, Ας ξεκινήσουμε, έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, λέω. Έχουμε μια καθυστέρηση 20 λεπτών περίπου. Δεύτερο πάνελ αφορά την σχέση αυτού του νέου μηχανισμού σας παρακαλώ πολύ, μήπως μπορούμε να κάνουμε λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε. Ε, μήπως θα μπορούσαν τα μέλη της γραμματείας να σταματήσουν τις συζητήσεις. Ωραία. Δεύτερο πάνελ για τη σχέση ανάμεσα στο νέο αυτό και την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Ίσως το παρατηρήσατε, στην σημερινή ακρόαση αλλάξαμε λίγο την ονομασία αυτού του ε, μηχανισμού. Στην πρόταση το όνομα ξεκινάει από το γράμμα N, την ε, γειτονία, ενώ εμείς αλλάξαμε λίγο τη σειρά εδώ και ξεκινάμε από το D που είναι η ανάπτυξη. DNICI, κανένας δεν αντέδρασε, θέλαμε να δώσουμε περισσότερη σημασία λοιπόν στην ανάπτυξη. Ε, ας δούμε λοιπόν τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη γειτονία τώρα. Πολύ δε περισσότερο που στην πρόταση την οποία λάβαμε, η θέση του Κοινοβουλίου γνώριθηκε πλήρως. Τι είχαμε πει εμείς, πρόσφατα μάλιστα, είχαμε πει ο μηχανισμός γειτονίας να παραμείνει χωριστός. Όπως επίσης και ο μηχανισμός για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγνοηθήκαμε πλήρως και θα αντιδράσουμε. Εγώ ως εισηγητής του Κοινοβουλίου θα αντιδράσω. Δεν τελείωσε αυτή η συζήτηση. Δεν δεχόμαστε αυτή την απόφαση που μας επιβλήθηκε. Επίσης, προτείνω να μειώσουμε λίγο το χρόνο που θα δώσουμε στους ομιλητές, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πέντε λεπτά λοιπόν σε καθένα από τους ομιλητές μας και θα είμαι και πολύ αυστηρός και με τους υπόλοιπους. Σκιώδεις ηγητές και λοιπούς. Έτσι ώστε στις 11.30 να ολοκληρώσουμε πρέπει να ψηφίσουμε για το βραβείο Ζαχάροφ στις 11.30. Αλλά ξεκινάμε λοιπόν με τον Αλεξέη Τζόνς, ε, ανώτερος, τέλεχος για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης της Αναπτυξιακής ε, Πολιτικής. Και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Σόνια Ρέινες Τζιβανίδη, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Συνδέσμου για την Οικοδόμηση της Ευρώπης. Αλέξη Τζόντς, σας δίνω το λόγο. Πέντε λεπτά δυστυχώς μόνο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να περιοριστώ στα πέντε λεπτά. Καταρχάς, λίγα λόγια για το EDCPM, που είναι, ε, είμαστε μια δεξαμενή σκέψη στο Μαστρίχτ. Ε, έχουμε και ένα μικρό γραφείο εδώ στις Βρυξέλλες και το βασικό καθήκον μας είναι να παρακολουθούμε και να συμβουλεύουμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής σε διάφορου τομείς όπως είναι η ανάπτυξη, το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και άλλου τομεί. Εγώ εργάζομαι πάνω στο ε, πρόγραμμα εξωτερικών υποθέσεων ε, της Ευρώπης και στο πλαίσιο αυτό αναλύουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, συμμετέχουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση των ε, προηγούμενων χρηματοδοτικών μέσων. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε τις ε, θέσεις μας ε, πάνω στο προτινόμενο μέσο γειτονίας ε, και ανάπτυξης και Θέλουμε να εξετάσουμε πώς αυτό το μέσο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιείται στη διεθνή σκηνή. Πράγματι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει διεθνής ε, παράγοντας, ε, κάτι που δεν θα γίνει όμως αποκλειστικά μέσω του μέσου αυτού. Το μέσο αποτελεί σημαντική πτυχή, δεν ε, θα αποτελέσει όμως τον μόνο τρόπο. Πολύ σύντομα, γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε, το παρόν πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εσωτερικά και εξωτερικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται να παραμείνει αξιόπιστη στο πολύ αστεθές ε, παγκόσμιο πλαίσιο όπου βλέπουμε νέες ε, τάσεις και δυναμικές ε, που προσφέρουν ε, μεν ευκαιρίες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις νέες καταστάσεις και να δράξει τις νέες ευκαιρίες που εμφανίζονται. Πράγματι και το θεματολόγιο 2030 αποτελεί σημαντική ευκαιρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει όσο γίνεται καλύτερα στο νέο αυτό θεματολόγιο. Και λοιπόν ε, στην ευρύτερη περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά κρίσεων και προκλήσεων ε, αλλά και εσωτερικά αμφισβητείται ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το Brexit και, το, και τη νέα κατάσταση στα κράτη-μέλη επίκυνται άλλωστε και ευρωπαϊκές εκλογές. Όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις στο μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να τονίσω δύο θέματα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματικός παράγοντας ε, στη διεθνή σκηνή, κάτι που κατά τη γνώμη μου ε, μπορεί να ε, εκφραστεί με δύο ερωτήματα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τη τη δυνατότητα να ενεργήσει ως μοχλός, να ανταποκριθεί σε ε, διεθνείς προκλήσεις και πώς μπορεί να συμφιλιώσει διάφορες αξίες και συμφέροντα. θα πρέπει να διασφαλίσει, να προστατεύσει τις αξίες της και να προωθήσει τα συμφέροντά της στις εξωτερικές δράσεις. Αυτά λοιπόν είναι δύο ερωτήματα που θα είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το νέο μέσο γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία ε, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Το επικροτούμε για διάφορου λόγου. Πρόκειται για πραγματικά πολύ τολμηρέ προτάσει που ε, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που ε, διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχάς βλέπουμε σημαντική αύξηση στον τομέα 6 που πλέον ε, δεν λέγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, σε διεθνές επίπεδο, αλλά στην ε, ε, γειτονική περιοχή και στο υπόλοιπο του κόσμου. Επικεντρωνόμαστε δηλαδή περισσότερο σε κάποιες περιοχές στις οποίες θέλει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξωτερικές της δράσεις. Είναι επίσης αρκετά ριζοσπαστικές οι προτάσεις αυτές στον τρόπο που προβλέπεται η απλούστευση και και η μεγαλύτερη ευελιξία στην δομή. Τονίζονται εδώ τρεις βασικοί πυλώνες ε, της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια, διεθνείς δράσεις και συμφέροντα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από το νέο αυτό μέσο. Ναι, δεν θα σας παρουσιάσω όλες τις διαφάνειες. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ερωτήματα που πιστεύουμε ότι θα είναι κρίσιμη συνεμασία και θα πρέπει να διασαφινιστούν ε, στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Καταρχάς, ε, αναφερθήκαμε στην ε, ευελιξία στο προηγούμενο πάνελ. Ναι, πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Δεν αρκεί από μόνο του όμως, δεν αποτελεί πανάκια θα πρέπει να εξετάσουμε τους κινδύνους ε, και τους ε, συμβιβασμούς που πρέπει να γίνουν ε, στο πλαίσιο της ευελιξίας. Επίσης, σήμερα το πρωί ακούσαμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι, πώς καταλαβαίνουν τα διάφορα θεσμικά όργανα την ευελιξία, διότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προωθηθεί αυτή η ιδέα και όσον αφορά τους απαραίτητους πόρους και όσον αφορά την προσαρμογή σε συνθήκες που συνεχώς αλλάζουν και την εξέβριση διαφορετικών εταίρων. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η ευελιξία θα πρέπει να θεσπίζεται στον κανονισμό, θα πρέπει όμως επίσης να διασφαλίζεται η ευελιξία στα επόμενα στάδια κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται η ευελιξία σε όλες τις διαδικασίες και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβάλλεται εις βάρος άλλων ε, πτυχών όπως είναι η παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγχος της και λοιπά. Κάτι που μπορεί να γίνεται εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία από τη μία και από την άλλη την προβλεψιμότητα και τη λογοδοσία. Επίσης ε, σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε οι εξωτερικές δράσεις να ε, ε, κατευθύνονται στρατηγικά. Σκοπός είναι να έχουμε πιο συνεκτική και στρατηγική εξωτερική δράση. Σας ανέφερα ότι το μέσο αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση αυτή της ιδέας. Ε, θα πρέπει όμως να έχουμε και ε, ε, στρατηγικό προσανατολισμό του μέσου αυτού. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Έχουμε κάποιες αφολίες όσον αφορά τα υπέρ και κατά του ring fencing και των εχεγγιών. Ίσως αυτός δεν είναι ο... Ίσως δεν είναι αυτές οι πιο βασικές αρχές που θα πρέπει να κατευθύνουν την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε και τον σχεδιασμό του όλου προγράμματο. Και επίση έχουμε τώρα ένα πρόγραμμα με παγκόσμια στρατηγική, έχουμε την αναθεωρημένη πολιτική γειτονία. Έχουμε λοιπόν το στρατηγικό πλαίσιο και σύντομα μπορεί να έχουμε αναλυτικό κανονισμό για να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη. Φαίνεται όμως να λείπει εδώ πέρα ένας κρίκος σχετικά με τον σχεδιασμό των εξωτερικών δράσεων, ώστε να έχουμε τα πλεονεκτήματα των συνεργειών ανάμεσα στους διάφορους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Θα κλείσω εδώ. Πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας μετά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόνια Ράιζη Ζιβανίδη. Παρακαλώ, περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να πάρω το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι η Έπλο είναι ένα, μια ανεξάρτητη πλατφόρμα 38 ΒΚΟ από 16 χώρες. Θα μιλήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα και θα, μιλήσω, θα αναφερθώ στο θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Το ζήτημα είναι τι είδου παίκτη θέλει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λαμβάνουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με θέματα ασφάλειας και ειρήνης. Ο προϋπολογισμός δείχνει τους στόχους που έχουμε και βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Θέλει να έχει καθοριστικό ρόλο εδώ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλές προκλήσεις και υπάρχει ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, τέρος, αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι θα μπορούσε να ε, βοηθήσει το πρέμα τη Ευρώπη να υπερισχύσει. Οι πολιτικοί προσπαθούν να δουν τι θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα για τους ε, πολίτες. Πολύ, πολύ, ε, δεν είναι σωστός ο τρόπος να καλλιεργούμε τους φόβους των ε, πολιτών ή να θυσιάζουμε τις μακρόπνοες διεργασίες το βωμό των βραχυχρόνιων. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν μια αίσθηση του ανήκειν. Οι ηγέτες θα πρέπει να μιλάνε ξεκάθαρα για όλα τα θέματα και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία νομική βάση για να προωθήσει την ειρήνη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, νομίζω ότι από τότε που η σοβιετική στρατηγική δημιουργήθηκε, είδαμε ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας. Το θέμα μας είναι τι θα πετύχει αυτή η επένδυση και τι θεωρία, θεωρία βρίσκεται από πίσω. Ε, εμείς αναφερθήκαμε στο θέμα της ανοικοδόμησης, της ε, ε, το, ε, το, της πρόθεσης των ικανοτήτων και της ασφάλειας. Και αυτός είναι ένας τομέας συνεργασίας. Υπάρχει και το πρόγραμμα για την ειρήνη και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που είναι σημαντικό κατά την άποψή μας θα δείτε ότι υπάρχει κάποια δορφή σε DST στην νέα, ε, στο νέο προτινόμενο κονδύλιο. Αυτό είναι ένας τομέας ε, που πραγματικά θα θέλαμε τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εξετάσει τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει. Ε, υπάρχουν θέματα που ε, φαίνεται να είναι ελκυστικά από πολιτική άποψη, αλλά πολύ συχνά απογοητεύουν. Υπάρχουν κυβερνήσεις που επένδυσαν δισεκατομμύρια σε αυτούς τους τομείς και το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Το, το... Η προσέγγιση μας ό,τι αφορά το πολιετές πλαίσιμο είναι ότι θα θέλαμε να μπορέσει να διαδραματίσει με μεγαλύτερο ε, ε, ειρηνευτικό ρόλο μας απασχολούν μακροπρόθεσμα τα θέματα της ανθρώπινας ασφάλειας. Την τελευταία φορά που ήρθα εδώ ασχοληθήκαμε με θέματα σταθερότητας, ειρήνης και χαιρόμαστε που τα χαρακτηριστικά ε, αυτά συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πρόταση και ιδιαίτερα το άρθρο 3 ε, γίνεται μία αναφορά σε μία σειρά από δράσεις ανεξάρτητα από την γεωγραφική θέση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί που εργάζονται επί αυτών των θεμάτων στη Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά την πρόταση NDICI, Είδαμε με χαρά μας ε, την αύξηση των κονδυλίων για εξωτερικές ε, δράσεις, συμπεριλαμβάνοντας μία αναφορά στην ειρήνη σε ένα γεωγραφικό πρόγραμμα, ε, έγινε αναφορά σε όλους τους πυλώνες, αλλά ε, μας απασχολεί το γεγονός ότι δεν είναι συγκεκριμένος αυτός ο στόχος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να μπει κατά μέρο αυτό το θέμα. Η ισότητα μεταξύ των δύο φίλων συζητήθηκε στα προηγούμενα πάνελ. Χαιρόμαστε που γίνεται αναφορά σε αυτό αλλά βεβαίως με μία, με και μοναδική αναφορά τα πράγματα δεν θα μπορέσουν ε, να πάρουν το δρόμο τους. Ε, είδαμε να γίνεται μία αναφορά στην πρόληψη των συγκρούσεων ε, και την αξιολόγηση της, του θέματος της ενσωμάτωσης της ένταξης των γυναικών. Υπάρχουν στοιχεία, ε, στοιχεία της SPSC που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παρατήματα της πρότασης και μας απασχολεί ότι υπάρχουν δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται. Έχουμε συγκεκριμένες τροπολογίες και δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το ρόλο της και το είδος της ασφάλειας που θέλει να επιτύχει. Πιστεύω, ε, η κυρία Μοργκερίνη είπε ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να ακολουθεί τις πολιτικές και το θέμα μας είναι πως θα έχουμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την πρόταση και με ανυπομονησία περιμένουμε συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους κοιότητες ηγητές. Οι συντηρητικοί δεν έχουν ορίσει κάποιον. Σαν και, σαν και ήταν εδώ αλλά έφυγε για τους πράσινους. Μισελ Ρεμόν. Εσύ αλλάξατε. Οκ, okay, κυρία Χάουταλα. Για τους πράσινους. Θα είμαι σύντομη. Επανέρχομαι στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε το πρώτο πάνελ. Για την συνεισφορά του μηχανισμού στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Χαίρομαι που η κυρία Ρέντ Ιβανίδη είπε πως το άρθρο 9 του CBSD είναι πολύ πιο λεπτομέρειες από οποιοδήποτε άλλο, κατά παράξενο τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό αυτή τη δράση θα ενισχύσετε την δημιουργία ικανοτήτων σε στρατιωτικούς φορείς. Αυτό αφορά η ασφάλεια. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε χάσει πλήρως την ιδέα της ανθρώπινης, της ατομικής ασφάλειας. Με αυτήν είχαμε ξεκινήσει όταν μιλούσαμε στον ΟΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς μπορούμε να την ξαναβάλουμε λοιπόν, να την ξαναεντάξουμε στο κάδρο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ για την Γκουέ, η κυρία Λέζινγκ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε από τους προσκεκλημένους μας και από την συνάδελφο την κυρία Χαουτάλα. Το θέμα είναι τι ρόλο θέλει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς, ε, Ποιο στρατηγικό στρατηγικός είναι ο σωστός και μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ακτιβιστή για την ειρήνη και πώς μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοιος. Νομίζω ότι οι περισσότερες στρατιωτικές επενδύσεις δεν θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ενώ στο, στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την, ε, για την άμυνα δεν ε, βλέπουμε σχεδόν καθόλου πολιτικά έργα, μη στρατιωτικά έργα. Να σας αναφέρω κάποια από αυτά που καταργήθηκαν. Η υποστήριξη των ε, των ε, παιδιών ε, σε ένοπλες ζώνες, ε, η επανένταξη γυναικών που συμμετείχαν, που συμμετείχαν σε ένοπλες σειράξεις κλπ. Τι μπορούμε συνάδελφοι να κάνουμε για να αντιστρέψουμε αυτή τη μεταφορά του βάρους και να έχουμε μέτρα οικοδόμησης της ειρήνης. Ο κ. Καστάλτο από την FTD δεν τον βλέπω εδώ. Έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Η κυρία Μακάβαν από του σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση προς τον κύριο Τζόουνς. Είπατε ότι... Νομίζω ότι είπατε, ξέρω ότι έπρεπε να βιαστείτε, αλλά είπατε Αναφερθήκατε στα εχέγγυα τα οποία μπορεί να είναι εις βάρος ε, της ευελιξίας. Ε, ναι, το καταλαβαίνω. Αν έχει κανείς υπερβολικά πολλούς ε, στόχους, Ε, πώς μπορούμε να μιλάμε για εταιρική σχέση αν εμείς επιβάλλουμε όλα τα μέτρα. Απ' την άλλη όμως πώς μπορεί να πετύχει κανείς τα εχέγγυα που θέλουν οι ευρωβουλευτές. Πώς μπορούμε δηλαδή να φροντίσουμε ότι θα ε, γίνεται σεβαστή η ισότητα των δύο φύλων, η προστασία του κλίματος κλπ. Ε, βλέπω ότι υπάρχει μια Πολωνέζα συνάδελφος που έχει αντικαταστήσει τον κύριο Κόρβι Μίκε. Σόσνεξ. Σόσ, σόσναξ. Δεν ξέρω αν διαβάζω καλά το όνομά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, ε, ε, ε, ε αποτροπή ένοπλων σειράξεων ε, με χρηματοδότηση. Τίποτα, τα χρήματα αυτά θα τα κλέψουν ε, οι διαθαρμένες κυβερνήσεις. Και μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε εδώ πέρα το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη με κάτι τέτοιο. Ισότητα ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για ισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ή μιλάμε για ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο. Σε κάθε οδηγία ε, του Κοινοβουλίου παραβιάζεται η αρχή αυτή μιλάμε για ειδικά δικαιώματα για τις γυναίκες. Δεν έχουμε ίση μεταχείριση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δικές μας χώρες, ίσως θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα την ισότητα. Οπότε έχετε ένα πρόβλημα με το Κοινοβούλιο, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε άλλη στιγμή. Δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, έχουμε καθυστερήσει. Ο λόγος ξανά στον Φέλιξ Φερνάντες Σο για τρία λεπτά. Ορισμένες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν μπορεί να τις απαντήσουν οι συνάδελφοι που δεν έλαβαν και το λόγο, ε, θα είναι πιο συγκεκριμένοι από μένα. Χίλτα Χάρτμαν, υπεύθυνη της ε, ε, υπηρεσία εξωτερικών οργάνων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία σχόλια. Η, ο τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσω της ειρήνης και της σταθερότητας, μέσω προσέγγισης του θέματος με μια αμοιβαία ωφέλιμη με ένα αμοιβαίο ωφέλιμο τρόπο. Ο στόχος ήταν πάντοτε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τα εργαλεία μας. Όπως είπαν και οι ομιλητές, το, ο μηχανισμός που έχουμε για την ειρήνη και την σταθερότητα αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί για να προληφθούν οι σειράξεις, να οικοδομηθεί η ειρήνη και ταυτόχρονα να προωθηθεί μια, ε, ένας ε, ε, πολυφωνικός τρόπος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ειρήνης. Πολυμερής τρόπος. Αυτά θα ενισχυθούν και στο μέλλον και ήδη συμπεριλαμβάνονται στις ε, υπερταχείες ικανότητες τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε στον αντίστοιχο πυλώνα και θα στηριχθούν με ένα προπολισμό 4 δισεκατομμυρίων. Θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν λοιπόν στο μέλλον. Δεύτερο σχόλιο μου, για τις συγκεκριμένε ερωτήσεις που έθεσαν κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με το ICSP. Ο στόχος θα διατηρηθεί. Το, ο μηχανισμός θα μεταφερθεί ως έχει στο NDICI, στο μηχανισμό ε, τον οποίο συζητούμε. Ένα κομμάτι μικρό θα πάει στην ε, ειρήνη, στο θεματικό πρόγραμμα και ένα κομμάτι στον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης, το μεγαλύτερο. Οι στόχοι όμως που διέπουν αυτή τη στιγμή το μηχανισμό για τη σταθερότητα και την ειρήνη θα μεταφερθούν 100% στο NDICI. Όμως για λόγους νομοτεχνικούς περιορίσαμε αυτή τη στιγμή την παρέμβασή μας. Δηλαδή δεν, αναφερόμαστε, δεν αναφέρουμε λέξη προς λέξη τους στόχους ε, για λόγους ε, νομοθετικής οικονομίας. Έχουν συμπεριληφθεί όλα όμως, παρόλο που δεν είναι λέξη προς λέξη. Πάντως είμαστε ανοιχτοί, αν θέλετε, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στον κοινωνικό μηχανισμό. Τρίτο μου σχόλιο. Πώς όλα αυτά σχετίζονται με άλλες δράσεις στήριξης της ειρήνης και της ε, σταθερότητας. Ο προϋπολογισμός της ε, εξωτερικής και πολιτικής πολιτικής ασφάλειας που δεν είναι τμήμα του NDICI θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί ή ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης θα καλύπτει αφενός το μηχανισμό Αθήνα και αφετέρου την ανάπτυξη ικανοτήτων που καλύπτονται από το μηχανισμό Αφρικανικής Ειρήνης, αλλά με ένα αντικείμενο πιο παγκόσμιο. Μαζί με λοιπόν με το NDICI αυτό τι μηχανισμοί θα διατηρήσουν και θα ενισχύσουν ότι υπάρχει ήδη και θα επιτρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο πιο πρωταγωνιστικό στην παγκόσμια ειρήνη με ένα πολυμερή τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Το λόγο τώρα με την Φεράνα, ε, Διευθυντή ε, Στρατηγική από τη Γενική Διεύθυνση Γειτονία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να εστιάσω την προσοχή μου περισσότερο στο θέμα της ε, γειτονίας. Τώρα, για να φερθώ στον όλο στόχο του μηχανισμού, πιστεύω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας διπλής πρόκλησης. Από τη μία πλευρά να υπάρχει μία δράση σε ό,τι αφορά τις γενικές προκλήσεις, αλλά χωρίς να αμπληθούν ε, οι πολιτικές μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό θέμα. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο συμπληρωματικά μέσα, ελαστικότητα από τη μία πλευρά και έγιναν πολλές συζητήσεις για το θέμα της ευελιξίας. Από την άλλη πλευρά προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των μεμονωμένων πολιτικών. Πιστεύω ότι έχουμε τρία στοιχεία στην πρότασή μας για την γειτονία. Πρώτο, να διατηρήσουμε τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής γειτονίας συμπεριλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών στο μηχανισμό. Και ένα και μηχανισμός δεν σημαίνει και μία πονιαία πολιτική. Αυτό θα έχει στόχο τη διατήρηση της διαφοροποιημένης προσέγγισης που είναι ένα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής γειτονίας. Θα συνεχίσουμε με τη συγκεκριμένη σχέση με τη χώρα, δημιουργώντας ε, εταιρικέ ε, ε, συμφωνίες, συμφωνίες σύνδεσης. Συνεπώς το πλαίσιο για την πολιτική παραμένει ως έχει. Αυτό που αλλάζει είναι το χώρο, το δοχείο μέσα στο οποίο σχεδιάζεται αυτό διατηρείται δικότητα σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις. Δηλαδή το αντίστοιχο του προγράμματος ομπρέλα παραμένει και επεκτείνεται και σε μερικά επιπρόσθετα κριτήρια για μετανάστευση, κινητικότητα, κράτος δικαίου και ε, οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να είναι κριτήρια ε, για να ανταμείβονται οι καλές επιδόσεις. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην πρόταση για αυτό το ε, μηχανισμό. Διακρατική, διασυνοριακή συνεργασία, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο δράσης σε ό,τι αφορά το παρόν μέσον δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό με την πρόταση του ε, μηχανισμού είναι αυτό που κερδίζουμε. Καταρχάς, ε, κερδίζουμε μία ασφάλεια σε ό,τι αφορά τα κονδύλια ε, και βεβαίως από την άλλη πλευρά ευελιξία και πρόσβαση σε αυτό το προστατευτικό μηχανισμό που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες κρίσεις. Αν κοιτάξουμε την κατάσταση στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία, αυτό αυτό θα είναι ένα διαχωριστικό για συγκεκριμένες πολιτικές γειτονίας, παράλληλα με έναν άλλο μηχανισμό προστασίας που θα παρέχει ευελιξία. Για να είναι βεβαίω αποτελεσματική η ευελιξία θα πρέπει να τη κάνει σωστής διαχείρισης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πώς θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να ακούσουμε τις, απόψεις, τις απόψεις σας έτσι ώστε να την κάνει καλής διαχείρισης αυτή η ευελιξία πάνω σε θεσμική βάση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε αυτή την πρόταση σαν κάτι που προσφέρει επιπλέον ευελιξία στην πολιτική γειτονία και ε, που δεν είδε την αμβλήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί λεπτά Φιλιμπέρτος εγκριγόνται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις της συναδέλφου σχετικά με το μέσο γειτονία και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ε, εισακούστηκε η θέση του Κοινοβουλίου και όσον αφορά τη γειτονία όμως και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο στόχος, τα ποσά, ο τρόπος εφαρμογής έχουν διατηρηθεί απολύτως και πιθανότατα να ενισχυθούν αν όλοι το επιθυμούμε. Νομίζω ότι στο προηγούμενο πάνελ ομιλητών ακούστηκε μία παρατήρηση σχετικά με τις ε, παρεμβάσεις ε, ε, υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι αυτές λείπουν από το νέο σχέδιο, αλλά όχι, αυτό δεν ισχύει. Όλα αυτά έχουν διατηρηθεί και μπορούν να εξεταστούν περαιτέρω. Μάλιστα, νομίζω ότι ανάμεσα στο προηγούμενο πάνελ και το τωρινό ακούστηκαν διάφορες παρατηρήσεις, για παράδειγμα ότι στον κανονισμό για το μέσο γειτονίας και ανάπτυξης έχουν αποδυναμωθεί κάποιες πτυχές, ενώ όσον αφορά την ασφάλεια είναι υπερβολικά αναλυτικό το μέσο. Έχουμε δώσει πληροφορίες στα κράτη-μέλη μας που δείχνουν τι υπήρχε στον ε, ισχύοντα κανονισμό και τι δεν έχει συμπεριληφθεί στον ε, κανονισμό για το μέσο γειτονία, ε, τον κανονισμό NDICI. Όλα αυτά βέβαια μπορούν πάντα να τροποποιηθούν με την επιφύλαξη που ανέφερα πριν, να μην έχουμε υπερβολικά αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τα άρθρα του κανονισμού. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω αυτό που το ECDPM ε, περιέγραψε ως ε, το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή να εξυπηρετούνται ε, διεθνείς στόχοι και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή είναι σημαντική η ε, ιδέα και δεν θα πρέπει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντίκυνται στους διεθνείς στόχους. Αντιθέτως, θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις συνέργειες που μπορούμε να εντοπίσουμε στο επίπεδο αυτό. Στον διασυνδεδεμένο κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα δεν βλέπουμε να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη διαχείριση πολύπλοκων φαινομένων όπως είναι η ε, αύξηση του πληθυσμού, η αστάθεια κλπ. Δεν βλέπουμε δηλαδή πώς μπορεί να είναι διαφορετικά τα συμφέροντα των ε, εταίρων μας από τα δικά μας. Το θεματολόγιο βιώσιμη ανάπτυξη ε, αποτελεί πλατφόρμα για να αναζητηθούν αυτά τα κοινά συμφέροντα. Κατά την εξέταση θεμάτων όμως όπως είναι η μετανάστευση, ε, και οι αιτίε τη αστάθειας νομίζω ότι έχουμε πολλά να μοιραστούμε με του εταίρου μας και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί με τόσο ανοιχτό τρόπο το μέσο αυτό. Μία τελευταία παρατήρηση σχετικά με τον προγραμματισμό. Ερμηνεύτηκε από το ECDPM ε, ως ε, το, τον κρίκο που λείπει, αλλά νομίζω ότι ε, σε διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας, σε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη μακροπρόθεσμη βοήθειά μας προς διάφορες χώρες και περιφέρειες του κόσμου και νομίζω ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του προγραμματισμού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, αλλά για δύο λεπτά. Δύο λεπτά, Αλεξέη Τζόνς. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Προτού απαντήσω στην, ερώτηση, στη συγκεκριμένη ερώτηση που τέθηκε ε, για τα εχέγγυα. Μια διευκρίνηση. Αυτός ο κρίκος που λείπει είναι ανάμεσα ε, στον ε, στο μέσο αυτό και τον προγραμματισμό. Θέλουμε δηλαδή να μεταφερθούμε από την αναπτυξιακή βοήθεια σε μια γενικότερη στρατηγική εξωτερική δράσης. Ανάμεσα λοιπόν στο πολιτικό πλαίσιο και στον προγραμματισμό ε, θα, γίνουν, ε, ε, θα ληφθούν κάποιες σημαντικές αποφάσεις και λείπει εδώ ο τρόπος λήψης των αποφάσεων αυτών. Η αναπτυξιακή βοήθεια πώς θα ταιριάξει και τι σχέση θα έχει με άλλους πυλώνες των εξωτερικών δράσεων. Εδώ κάτι λείπει λοιπόν και γεωγραφικά και θεματικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική για το θεματολόγιο 2030. Θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε περαιτέρω ε, προσανατολισμό για το πώς ε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα θέματα αυτά. Όσον αφορά ε, την διάθεση πιστώσεων και τα εχέγγυα, θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο τι υπάρχει στον κανονισμό και στο τι θα πρέπει να ελέγχεται εκ των υστέρων. Θα πρέπει να υπάρχει διαφανής τρόπος να δει κανείς πώς έχει δαπανίσει τους σπόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι τα εχέγγυα ε, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο όχι του κανονισμού, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν σε άλλο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ήθελα να πω ότι είναι υπερβολικά αναλυτικές ε, οι προτάσεις. Στον προϋπολογισμό έχουμε υπερβολικά... Στον προϋπολογισμό τονίζεται υπερβολικά η πτυχή της ασφάλειας. Δεν λέμε ότι η ασφάλεια δεν είναι σημαντική. Λέμε όμως ε, ότι έχουμε επενδύσει υψηλού κινδύνου ε, στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη, για παράδειγμα, και δεν ξέρουμε πώς θα ληφθούν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θέλαμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να ε, εντείνει τον ρόλο του στην εξέταση των θεμάτων αυτών, διότι η κοινωνία των πολιτών θα εξετάσει τη λειτουργία των ε, θεμάτων ε, αυτών με βάση το παρελθόν. Και θα δείτε και στο Αφγανιστάν και αλλού ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε δεν ήταν πολύ αποτελεσματική. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν προτείνονται κάποια ε, πολιτικά μέσα εδώ, εγώ θα ήθελα το Κοινοβούλιο να ζητήσει αλλαγή της ονομασίας αν μη τι άλλο για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Euh, euh, ευχαριστώ για τρία λεπτά ο Αντώνιο Πατσέρη. Ευχαριστώ Κρίστιαν. Βεβαίω και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αφιτρίωνε. Θα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που εκφράστηκαν θα ήθελα να, στήσω, να στείλω δύο βασικά μηνύματα και ελπίζω να είμαι σαφής. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι η ευελιξία αυτή καθ' αυτή δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ένα θετικό τρόπο προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η δράση της Ένωσης και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να οριστούν καλύτερα οι λεπτομέρειες. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί και με λάθος τρόπο, γιατί αν υπάρξει πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια της ε, Επιτροπής, πέρα από τον προγραμματισμό που έχει γίνει, θα ανακύψει ένα πρόβλημα. Το δεύτερο μήνυμα. Γίνεται μία συζήτηση σχετικά με το ενιαίο μηχανισμό. Ο στόχος των τετσάρων συνεισηγητών ήταν να δώσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία εργασία που θα βασίζεται σε αυτό το πρόγραμμα του ενιαίου μηχανισμού που προτείνεται από την Επιτροπή. Μετά θα ξεκινήσει μια φάση συζητήσεων και τροπολογιών. Εγώ απλά και μόνο θα ήθελα να πω και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι η θετική κατάληξη αυτής της συζήτησης θα συνδέεται στενά με την επίτευξη ενός μεγαλύτερου, μιας μεγαλύτερης δυνατότητας ελέγχου και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για όλα αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σε ένα εργαστήριο με την ΑΦΕΡ και την ΤΕΒΕ στις 15 Οκτωβρίου και θα δούμε διεξογικότερα τα θέματα καταβάλλοντας μια προσπάθεια με το τέλος του Οκτωβρίου να υποβάλουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ευχαριστώ, Λίντα Μακάθιν. Παρακαλώ, τις τελικές παρατηρήσεις. Θέλω μόνο να πω ότι ο χρόνος μας πιέζει σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αυτής της νομοθεσίας. Οι συνάδελφοι δουλεύουν πολύ σκληρά. Είναι το πιο σημαντικό θέμα το οποίο θα χειριστούμε μέχρι τις εκλογές. Καλό, καλύτερο είναι να πετύχουμε το ευέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ τους προσκαλεσμένους μας.